Um, Ως Σουηδέζα θα μπορούσα να πω ένα ε, επιπρόσθετο ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και σας ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης για τις απαντήσεις σας. Τώρα έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για ε, μια καταληκτική δήλωση πέντε λεπτά πριν λήξει και η συνεδρίασή μας. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. So, uh, honorable members of uh, Parliament. κύριε Ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ευκαιρία για ε, αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τον μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που με υποβάλλατε που και που καταλαβαίνω θα απαιτήσουν περαιτέρω δουλειά και παρακολούθηση. Πάντως είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ στενά με το Ευρωκοινοβούλιο καθώς και εγώ ίδιος ε, έχω διατελέσει ευρωβουλευτής για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω ότι σας οφείλω μια, απάντηση για μια ερώτηση που τέθη και με επικρίνατε που δεν μπόρεσα μέσα σε δύο λεπτά να την απαντήσω και αφορούσε τα ασφάλματα τα οποία έγιναν στην Λετωνία ε, κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της κρίσης και νομίζω πως μπορείτε να βρείτε κάποιες απαντήσεις στις ειδικές συστάσεις προς τη Λετωνία. Υπάρχουν διάφορες συστάσεις πολιτικής όσον αφορά την ενίσχυση της ανεξαρτησίας μας στην ενέργεια. Πολύ σημαντικό θέμα σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο. Στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στα εισοδήματα συμπεριλαμβανομένων ε, των αλλαγών ε, στη συνεφορολογική πολιτική, ενίσχυση του δικαστικού σώματος, αντιμετώπιση προβλημάτων αφαιρεγγιότητας, Διάφορες λοιπόν συστάσεις ε, για τη χώρα μας που λάβαμε και που ε, εντόπισαν προβλήματα τα οποία ε, θα έπρεπε η Λετωνία να αντιμετωπίσει. Ελπίζω πως η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί τώρα, γιατί πριν δύο μέρες μόλις κάναμε, είχαμε εκλογές, ε, Ελπίζω λοιπόν ότι θα δεχτεί και θα λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις συστάσεις η νέα κυβέρνηση και θα μπορέσει έτσι να αντιμετωπίσει τις πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Λετωνία. Όσον αφορά την εργασία της νέας Επιτροπής, θα πρέπει και να τονίσω για μια ακόμη φορά πως πρόκειται για μια νέα δομή, οπότε δεν έχουν όλα κουρδιστεί στην τελευταία λεπτομέρεια, αλλά μπορώ σαφώς να σας πω ότι όλοι οι υποψήφοι επίτροποι με τους οποίους έχω συνομιλήσει διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, είναι πρόθυμοι για να εργαστούν ομαδικά, ε, οφείλω μου τους ή άλλως να δουλέψουμε ομαδικά ακόμα και αν ε, προερχόμαστε από διαφορετικά πολιτικά ε, κόμματα, ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να αποδώσουμε ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα θέματα που ανησυχούν τον κόσμο. Τα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης, τα θέματα της απασχόλησης, της εξέλιξης των μισθών, τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για αυτή την ακρόαση και πραγματικά προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί σας και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Just a few remarks on the... Μερικές παρατηρήσει για την διαδικασία που θα ακολουθήσει. Θα γίνει κοινή αξιολόγηση, συνεδρίαση αξιολόγηση με τους Προέδρους των δύο Επιτροπών και τους συντονιστέ. Θα γίνει στις 7 ε, απόψε στην αίθουσα 3G2 στο κτίριο ASP. Θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη τις διάφορες ε, ανησυχίες ε, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ε, επιστολής αξιολόγησης και που θα κυκλοφορήσει αργότερα απόψε. Η προθεσμία για σχόλια για την επιστολή είναι πρωινή, αύριο στις 7 Οκτωβρίου δηλαδή, και οι συντονιστές είναι οι, οι άνθρωποι επαφής και ζητώ από τους συντονιστές ε, της Επιτροπής Απασχόλησης να έρθουν εδώ κοντά μου για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε τώρα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Οι συντονιστές λοιπόν ε, της Επιτροπής Απασχόλησης παρακαλώ ελάτε εδώ κοντά μου στο Προεδρείο. Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά κύριε Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ όλα τα μέλη των δύο επιτροπών που ήσασταν σήμερα εδώ και που θέσατε ε, ευφυείς ερωτήσεις.